Κυρίε και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασής μας. Πρώτο θέμα της σημερινής σας διάταξης αφορά βεβαίως ε, το πρόγραμμα ε, τη σημερινή συνεδρίασης στη μέση διάταξη υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, όχι από ό,τι βλέπω, οπότε εγκρίνεται. Έχω και ένα καθήκον να εκτελέσω. Η γραμματεία της Επιτροπής ΠΕΤΗ στη γραμματεία μάλλον εργάζεται ο κύριος Άλντερς Έντερς, ο οποίος ε, συνταξιοδοτείται μετά από 30 χρόνια εξαιρετική συμβολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξ αυτών ε, πέρασε 25 χρόνια σε διάφορα όργανα, θεσμικά. Τα τελευταία 5 χρόνια ήταν, ήταν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εργάστηκε επί αναλύσεων, μελετών κτλ. Εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής Αναφορών θα θέλαμε να ευχηθούμε στον κύριο Άντερσον ό,τι καλύτερο. Η συνεργασία μαζί του ήταν πολύ σημαντική και είναι χρέος μας να του εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όλα όσα έκανε. Και περνάμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνέταξε έκθεση με θέμα την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον κύριο Λεομπρίνκατ που είναι εισηγητής, συντάκτης της έκθεσης αυτής. Θα του δώσουμε το λόγο να ακούσουμε την ε, ε, παρουσίασή του και στη συνέχεια θα δώσει το λόγο στους ε, συντονιστές και στους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Ε, καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση που σας παρουσιάζουμε σήμερα ε, ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα απαλλαγή για τον Γενικό ε, Προπολογισμό του 2014. Σχετικά με το αν το, η Κομισιόν έχει αξιοποιήσει ορθά τις αρμοδιότητε τη όσον αφορά την υποστήριξη και τον έλεγχο των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του ενουσιακού δικαίου. Λόγω του ότι η εποπτεία της Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη είναι περίπλοκο ζήτημα, καθώς καλύπτει πολλούς ε, οριζόντιους τομείς πολιτικής, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην έκθεση αυτή σε ορισμένα πραγματικά στοιχεία. Στο, στη διαδικασία αυτή μιλήσαμε με πολλούς εμπλεκόμενους. Την κυρία ε, Βίξτρομ, την πρόεδρο της ε, Επιτροπής ΠΕΤΗ και θέλω να την ευχαριστήσω για το γεγονός ότι η ίδια απεδέχθη να είναι ε, ομιλήτρια σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώσαμε το, ε, στις 24 Σεπτεμβρίου. Συζητήσαμε και με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ε, ως ε, επίσης εμπλεκόμενη στην, ε, στο ζήτημα της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας. Γιατί το κάναμε αυτό, διότι ε, επικεντρωθήκαμε ακριβώς σε εσά και στην Ευρωπαία Δημοσιολαβήτρια ακριβώ γιατί το έργο σας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες της Ένωσης και αναγνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών, μέσω των αναφορών που επεξεργάζεται, μας παρέχει σημαντικότατες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το δίκαιο εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεσή μας ε, επικεντρωθήκαμε σε μια πολύ σημαντική ε, διάσταση αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις εποπτικές δραστηριότητες της Κομισιόν που είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά την πρόληψη, την ανείχνευση και τη διόρθωση παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πολύ συχνά η Κομισιόν χρησιμοποιεί τον όρο παρακολούθηση τη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Εμείς ε, λοιπόν καταλήξαμε σε μια ανάλυση του νομικού τοπίου της Ευρωπαϊκής Ένωση και των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, και έτσι η ομάδα μας λοιπόν μίλησε με μια σειρά από γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν αλλά και εκπροσώπους, με εκπροσώπους των κρατών μελών, έκανε συνεντεύξεις με πολύ σημαντικούς εμπλεκόμενους φόρους, θεσμικούς, επανεξέτασε διάφορες εκθέσεις που έχει συντάξει η Κομισιόν και εκθέσεις βεβαίως του ίδιου του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, αλλά και των ε, ανώτατων αρχών των κρατών μελών. Η εποπτεία της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου είναι εγγενώς ε, δύσκολο έργο. Και αυτό διότι το ενωσιακό δίκαιο είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Στην έκθεσή μας επισημαίνουμε τρει διαστάσει. Πρώτον, ότι υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλές νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής που πρέπει να παρακολουθηθούν. Δεύτερον, ότι οι τομεί αυτοί παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Και τρίτον, ότι ε, κάθε κράτο μέλο εφαρμόζει το νοσιακό δίκαιο με διαφορετικό τρόπο. Ε, πράγματι, η πρόταση της Επιτροπής Αναφορών να ενισχυθεί η κατάρτιση για την βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των ε, εθνικών αρχών για την ενίσχυση του, των δικαιωμάτων των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ε, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και εμείς. Εμείς λοιπόν ε, ε καταλήξαμε σε, σε δύο βασικά ζητήματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και εσάς είναι το δεύτερο και το έκτο σημείο. Πρώτον, ενθάρρυνση πολιτών στην παρακολούθηση και την ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων, την άσκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και ε, υποβολή εκθέσεων ετησίως σχετικά με την, με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου ε, περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητε που βεβαίως είναι και χρονοβόρες, χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη. Οι γενικές διευθύνσεις προσδιορίζουν πιθανές παραβιάσεις με τρεις τρόπους κατά κύριο λόγο. Πρώτον, ελέγχοντας τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ε, ε, οδηγιών, εξετάζοντας καταγγελίες αλλά και ε, διενεργώντας δικές τους έρευνες. Όσον αφορά ε, ε, τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, η Κομισιόν λαμβάνει 3 με 4 χιλιάδες νέες καταγγελίες κάθε χρόνο ε, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αριθμό των ερευνών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των διαδικασιών επί παραβάση ε, ανέρχονται σε περίπου χίλιε κάθε χρόνο. Οι περισσότερε παραβιάσει αφορούν κυρίω την καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και όχι καταγγελίε. Εκεί μιλάμε για περίπου 60 με 80% ανάλογα με το χρόνο βεβαίω. Υπάρχει μια διακύμανση. Μόνο μία από κάθε έξι ή 7 καταγγελίε τελικά ερευνώνται και αυτό γίνεται διότι μια συγκεκριμένη γενική διεύθυνση ε, μπορεί να έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει παραβίαση, δεν υπήρξε παραβίαση ή ότι υπάρχουν άλλες τρόποι για τη διόρθωση της παραβίασης πέραν της διαδικασίας επί παραβάση. Αυτό σημαίνει ότι πολύ λιγότερες περιπτώσεις τελικά ερευνώνται από όσες καταγγέλλονται. Στη βάση ε, των ερευνών που κάνουν οι ίδιες οι γενικές διευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ γενικών διευθύνσεων. Οι γενικές διευθύνσεις ε, προσδιορίζουν πιθανές παραβιάσεις μέσω άσκησης των ερευνητικών τους αρμοδιοτήτων. Ε, βάση επίσης ελέγχων καταλληλότητας άλλων ε, αξιολογητικών διαδικασιών που διενεργούνται. Βεβαίως αναφορές στον τύπο ή εκθέσεις από οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές ερευνητικές αρχές ή ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών. Και αυτές μπορούν να αποτελέσουν πολλές φορές πηγή. Η συνολική διάρκεια επίσης αυτών των ερευνών ε, είναι επίσης ένα ζήτημα. Ιδίως εκείνες που καταλήγουν τελικά σε διαδικασία παραβάση. Διαπιστώνουμε ότι κατά μέσο όρο χρειάζονται τρία χρόνια για να επιληθεί μια υπόθεση και περίπου 70 εβδομάδες ε, πολλές φορές ε, ε, δαπανώνται σε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πιλωτικές έρευνες που γίνονται εδώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξοικονομηθεί χρόνος στις διαδικασίες επιπαραβάση. Πρέπει να υπάρξει ιεράρχηση και σε τελική ανάλυση σε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις επιβάλλονται κυρώσεις ή πρόστιμα. Παρ' όλα αυτά, οι γενικές διευθύνσει και τα κράτη-μέλη αναφέρουν ότι η διαδικασία επιβαραβάση ε, αποτελεί ένα σχετικά αποτελεσματικό εργαλείο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το νησιακό δίκαιο παρά την διάρκεια, την πολύ μεγάλη διάρκεια, αλλά και τους πόρους που απαιτούνται. Η Κομισιόν επίση χρησιμοποιεί μια σειρά από εργαλεία για την προώθηση της συμμόρφωσης. Υπάρχουν καταυθυντήρε γραμμέ, για παράδειγμα, όσον αφορά την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, που χρησιμοποιούνται και αναγνωρίζονται ως αξία από τα κράτη-μέλη. Και θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί. Από την άλλη μεριά, ε, τα σχέδια εφαρμογής ε, για την, ε, για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων δεν χρησιμοποιούνται, παρά μόνο σπάνια. Χρειάζεται επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διαφάνεια. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι καταγγέλλοντες, τα κράτη-μέλη ε, τα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινό έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες που δυστυχώς πολύ συχνά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Στην έκθεσή μας περιγράφουμε τους κύριους τρόπους με τους οποίους η Κομισιόν επικοινωνεί με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Το αν οι πληροφορίε αυτές ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εμπλεκομένων φορέων ή αν θα μπορούσε να ε, ή ε, το αν δεν το κάνει είναι ένα βασικό ζήτημα που μας απασχολεί. Σίγουρα πάντως υπάρχει ένα χάσμα όσον αφορά τις προσδοκίες. Τηρώντας ενήμερους λοιπόν τους πολίτες, η Επιτροπή ΠΕΤΗ καταβάλει σημαντικότατες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και έτσι συμβάλλει στην κάλυψη του χάσματος, του χάσματος που σας περιέγραψα μόλις. Στο τέλος αυτής της έκθεσής μας για το τοπίο προσδιορίζουμε και μια σειρά από ευκαιρίες για την ενίσχυση της εποπτείας. Τρεις από αυτές αφορούν την ενίσχυση της διαχείρισης των ικανοτήτων, ιδίως την ε, διαθεσιμότητα συνολικότερων πληροφοριών όσον αφορά το χειρισμό των διαφορών υποθέσεων. Και ολοκληρώνουμε την έκθεσή μας αναδεικνύοντας την, ε, τις δυνατότητες που έχει το ελληνικό συνέδριο για τη διενέργεια ελέγχων σε αυτό το τομέα αναδεικνύουμε ε, ότι μπορούμε, για παράδειγμα, να εξετάσουμε μια σειρά από διαστάσεις ή μπορούμε να ε, πιέσουμε ε, και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη χρήση του ευρωνοσιακού προϋπολογισμού. Η διαχείριση των διαφόρων σταδίων των διαδικασιών για την επεξεργασία καταγγελιών επίσης είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως ε, είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρινκάτ για την παρουσίαση αυτή, για τις, παρουσ... για τις πληροφορίες που μας ε, δώσατε. Το ζήτημα αυτό βεβαίως μπορεί κανείς να το επεξεργαστεί πολλή πλευρά και με διάφορους τρόπους Βεβαίως προσπαθήσατε να μας δώσετε μια σαφή εικόνα, τα πράγματα όμως γνωρίζουμε ότι είναι πολύ περίπλοκα. Η Ευρωπαϊκή Πετροπή έχει πλέον πάρα πολλές αρμοδιότητες. Έχουμε μαζί μας και εκπροσώπους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους οποίους θα ήθελα να δώσω το λόγο για να τοποθετηθούν και εκείνοι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. honorable members. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Επίσης, ευχαριστούμε και τους συντάκτες της παρουσίασης για την συνεργασία όπως είχατε την δυνατότητα να αναφέρετε στις 24 Σεπτεμβρίου η παρουσία της Επιτρόπου. Όλοι εμείς καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον του ελεκτικού συνεδρίου σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της εφαρμογής του ενωσιακού νόμου. Είναι πολύ σημαντική η περιγραφή που κάνατε. Για πρώτη φορά μας δίνετε μια καλή ιδέα του πόσο τα εμπλεκόμενα μέρη ή τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη που συνεργαζόμαστε, τα κράτη-μέλη, πώς καταλαβαίνουν, κατανοούν όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή τους, ούτως ώστε να εφαρμόζουν έγκαιρα και σωστά τον ενωσιακό νόμο. Επίσης, αναγνωρίζετε όλες τις πολυπλοκότητες που αφορούν το ζήτημα αυτό. Κάποια από τα ευρήματά σας θεωρώ ότι περιλαμβάνονται στην πολιτική του 2017 της Κομισιόν. Έχετε όμως μια σειρά από προτάσεις τις οποίες θα προωθήσουμε μεταξύ των οποίων και η διευκρίνηση του πεδίου δράσης μας. Θέλουμε να, έχουμε, να είμαστε λίγο πιο έμπειροι με την ε, πολιτική αυτή. Χρειάζονται κάποια χρόνια από το 2016 που ξεκίνησε, το ώστε να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Έχετε και μια πολύ χρήσιμη ανάλυση των ε, λεγόμενων εργαλείων συμμόρφωσης, εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε από κοινού μαζί με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα και πότε, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται με έναν έξυπνο τρόπο ώστε να βοηθούν τα κρατημέλη να εφαρμόζουν τον ενωσιακό νόμο η διαφάνεια Επίσης τα ευρήματα του ελεκτικού συνεδρίου όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημεία που από κοινού μας με τα κράτη-μέλη μπορούμε να κάνουμε πρόοδο. Η αναφορά σας σημειώνει ότι οι ετήσιες αναφορές είναι καλής ποιότητας, υπάρχει όμως περιθώριο βελτίωσης και αυτό το σημείο θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Επίσης πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν και αυτά το ρόλο τους, μπορούν να είναι και τα κράτη-μέλη με τη σειρά τους πιο διαφανή σε ό,τι αφορά την μεταβίβαση του νοσιακού νόμου σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η αρχική μου αντίδραση. Θα εξετάσουμε από κοινού πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τα εργαλεία εφαρμογής, αλλά και να αυξήσουμε την ε, διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόλντες. Ο κύριος Τίμερμανς, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει πολύ συχνά ότι θα επιδείξουμε πυγμή και αποφασιστικότητα. Τέσσερις φορές το έχω ακούσει τουλάχιστον από τον κύριο Τίμερμαν. Εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το δίκαιο έχει αξία μόνο σε περίπτωση που πραγματικά εφαρμόζεται. Αλλιώς είναι καινογράμμα. Ο κύριος Γιάρα. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση γιατί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών ε, μπορώ να σας πω ότι είμαστε και κάτι σαν σεισμογράφος του ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θετικό μαντάτο είναι ότι οι πολίτες όχι μόνο δέχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως εξ αυτού ε, πηγάζουν και ορισμένες ε, προσδοκίες των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που σχετίζεται και με την εν γέννη ηθαγένεια του, του, του, του Ευρωπαίου πολίτη. Υπάρχουν λοιπόν αρμοδιότητες, ε, αυτό βεβαίως γι' αυτό δεν φταίτε εσεί, για το ποιοι τομεί τέλο πάντων αρμοδιότητα έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιου έχουν κρατήσει τα κράτη-μέλη περιγράφεται ότι επί της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ακόμα οδηγίες και κανονισμούς ως βασικό μέσο ε, θέσπισης νομοθεσίας. Και οι οδηγίες ιδίως ε, βεβαίως δίνουν μια πολύ μεγάλη πυκλομορφία ε, στα κράτη-μέλη όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής τους. Έχω λοιπόν να κάνω κάποιες να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, Ιδίως στον τομέα της, ε, του περιβάλλοντος. Πολλές φορές λαμβάνουμε αναφορές ότι δεν έχουν γίνει σωστές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι δεν τηρήθηκαν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, προστασίας της φύσης. Και εδώ, στην Επιτροπή ε, Πέτη, πολλές φορές λαμβάνουμε σε αυτούς τους τομείς την απάντηση από την Κομισιόν, ότι εμείς θεωρούμε δεδομένο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία με τον κατάλληλο τρόπο. Ε, εδώ θα θέλαμε η Κομισιόν να ασκεί μεγαλύτερη εποπτεία και στην διαδικασία του σχεδιασμού των έργων. Πολλές φορές υπάρχουν, για παράδειγμα, κατασκευαστικά έργα τα οποία ε, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και στη συνέχεια διαπιστώνεται, στο τέλος αφού ολοκληρωθούν δηλαδή, ότι δεν τηρήθηκαν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές. Ε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εδώ θα έπρεπε η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη τη Κομισιόν προ τα κράτη-μέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, δεν θα έβλαπτε κανέναν αν η Κομισιόν παρακολουθούσε τι διαδικασίε αυτέ εξ αρχή. Δεύτερο θέμα. Διαφάνεια. Σα υποστηρίζω πλήρω αυτά που είπατε. Αλλά έχω και ένα ερώτημα προς το ελεγκτικό συνέδριο. Τι ε, αίσθηση έχετε αποκομίσει από, την, από το έργο σας. Ξέρετε, οι νόμοι δεν πέφτουν από τον ουρανό. Η θέσπιση του ενωσιακού δικαίου είναι πραγματοποιείται μέσω μιας ε, περίπλοκης μεν αλλά απολύτως λογικής και προβλεπόμενης διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν το, τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμάς Ξέρετε, μας ενοχλεί πολύ συχνά το ότι αφού θεσπιστεί νομοθεσία, τα κράτη-μέλη συμπεριφέρονται σαν να μην συμμετείχαν ε, στη θέσπιση αυτής της νομοθεσίας και το, την ίδια στάση τηρούν και στη φάση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η προθυμία των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εσείς τι αίσθηση έχετε Υπάρχει διαφορά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, υπάρχει απροθυμία, υπάρχει προθυμία για την ε, εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Και ε, ερώτημα που συνδέεται με αυτό. Μήπως χρειαζόμαστε έναν σοβαρότερο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Να πάρουμε το παράδειγμα ε, τη γεωργική πολιτική. Εκεί τα πράγματα είναι άψογα δεν υπάρχουν προβλήματα, εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Γιατί όμως, διότι και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης είναι αυστηρότατες. Μήπως λοιπόν το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι οι αναφορές μας, ε, πρέπει να σας πω εγώ από τη δική μας πλευρά, ότι πάντοτε κατατείνουν σε αυτό, στο πώς θα εξασφαλιστεί η εφαρμογή της ε, νομοθεσίας. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες που έχουμε στα χέρια μας. Ο κύριος Όλης. For, uh, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ε, τους συντάκτες της εξαιρετικής αυτής αναφοράς που πραγματεύεται πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε για την εφαρμογή των ενωσιακών νόμων. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε διαφορετικά επίπεδα, σε πολλές περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ακόμη αρκετοί τομείς στις οποίες οι οδηγίες δεν εφαρμόζονται εγκαίρως και σωστά. Και υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Από την άλλη μεριά, ιδίως μετά την τελευταία οικονομική κρίση του 2004, αλλά και την εισχώρηση χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αναγκάστηκαν οι χώρες αυτές να μεταγράψουν την ενωσιακή νομοθεσία στις εθνικές τους νομοθεσίες κυριολεκτικά λέξη προς λέξη, κάτι το οποίο δημιούργησε χάος την εγχώρια νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις η εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας με την εγχώρια νομοθεσία ήταν προβληματικό. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι αναφερόμαστε στην συμμόρφωση, θα πρέπει να κρατάμε κατά νου ότι η συμμόρφωση δεν σημαίνει απαραίτητα μετάφραση κατά λέξη στην εθνική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε το πνεύμα και τη λογική της κάθε οδηγίας, σεβόμενη πάντοτε το εγχώριο νομικό πλαίσιο. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να αναφέρω από τη μία έχουμε την εφαρμογή, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργούν άριστες συνθήκες αξιολόγησης, αξιολογήσεις αντικτύπου της λεγόμενης των οδηγιών του ενωσιακού νόμου. Μπορούμε να συζητάμε την εφαρμογή, μπορούμε να συζητάμε την χρήση των οδηγιών, θα πρέπει όμως να συζητάμε και τον αντίκτυπο που έχει η ενωσιακή νομοθεσία. Σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικό να έχουμε έγκαιρη αξιολόγηση αλλά και να μπορούμε να έχουμε προτάσεις και τροπολογίες ούτως ώστε να έχουμε το περιθώριο να βελτιώνουμε τα αποτελέσματα και το νομικό πλαίσιο που προτείνουμε ούτω ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Από τη μία μεριά μπορούμε να έχουμε τις βασικές αρχές της νομοθεσίας και από την άλλη μεριά έχουμε και τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις και είναι ανάγκη να αξιολογούμε και τα δύο πράγματα. Από τη μία την αξιολόγηση και από την άλλη τον αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή των νόμων αυτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Όχι δίνουμε το λόγο σε εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ επικοδηματικές ε, οι παρατηρήσεις σας και ενδιαφέρουσες. Ξέρετε ότι βασικός στόχος της μελέτης μας ήταν να αξιολογήσουμε τη διαδικασία εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη-μέλη. Θα απαντήσω λοιπόν γενικά αλλά και συγκεκριμένα αυτό ποικίλει, γιατί εξαρτάται από το, από το είδος της νομοθεσίας, από την ε, περιπλοκότητα των, νομικών, νομικών μέσων, τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα πολιτικές, πολιτικής. Ορθώς ε, είπε και ο συνάδελφος ότι για πράγματα τα πράγματα είναι πολύ πιο προβληματικά στον περιβαλλοντικό τομέα. Υπάρχουν επίσης, υπάρχει επίσης η διάσταση των ε, εργαλείων και των μέσων που έχουν στη διάθεση τα κράτη-μέλη και οι διοικητικέ τους ικανότητες. Κάθε νομική πράξη λοιπόν παρουσιάζει συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της από την πλευρά των κρατών μελών. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σημαντικέ διαφορές σχετικά με τις, ε, τους συνταγματικούς, νομικούς και πολιτικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε ε, χώρα. Οι βασικές προκλήσεις, αφού θέλετε να συνοψίσω, είναι ότι παρά το γεγονός ότι κάθε νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει συγκεκριμένες, ε, δυσκολίες, θα πρέπει πιο γρήγορα οι ίδιε οι διοίκησει να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τα προβλήματά τους, τι καθυστερήσει, καθώ και τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτά. Πρέπει να μειωθούν οι καθυστερήσει, πρέπει να δούμε αν η εφαρμογή βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχουν οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και αν οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με το ίδιο το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν οι κεντρικές κυβερνήσεις αξιοποιούν αποτελεσματικά το περιθώριο που δίνει κάθε οδηγία. Και πρέπει επίσης να εξετάσουμε τον ίδιο το ρόλο της Κομισιόν ως παράγοντα διευκόλυνσης που παραμένει κεντρικός. Πολλές φορές το ερώτημα που μας απευθύνεται είναι πού είναι το βασικό πρόβλημα, στα κράτη-μέλη ή στην Κομισιόν. Εμείς, ξέρετε, προσπαθήσαμε να ε, να αποτυπώσουμε ένα στιγμιότυπο αν θέλετε ε, για να δούμε πού ακριβώς ε, πρέπει τελικά να γίνουν προσπάθειες. Βεβαίως το βασικότερη αρμοδιότητα, η βασικότερη ευθύνη ε, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, για να μπορέσει να εφαρμόσει τις επιπτωτικές δραστηριότητε. Ευθύνη όμως έχουν και τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό εγώ ε, βασίζομαι στη δική σας επιτροπή, στους εμπλεκόμενους, στους ίδιους τους πολίτες. Διότι ε, η διαφάνεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Πρέπει να έχουμε βεβαίως υπόψη μας τις προσδοκίες ε, που έχουν οι πολίτες μας. Πρέπει γι' αυτό να αναπτυχθούν νέοι μηχανισμοί και από αυτή την άποψη χαιρετίζω και τα σημερινά σχόλια της Κομισιόν που μας είπε ότι θέλει να ενισχύσει τα εποπτικά της εργαλεία και ε, συμφώνησε με, την, ε, με το βασικό πόρισμα της δικής μας μελέτης ότι θα πρέπει οι νέοι μηχανισμοί να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ευθύνες που υπάρχουν σε επίπεδο κομισιών και κρατών μελών. Πιστεύω λοιπόν ότι μια διάσταση που πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχέστερα είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επαρκής έμφαση στους ανθρώπινους πόρους που είναι διαθέσιμοι καθώς η κάθε γενική διεύθυνση λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Η πλειονότητα του προσωπικού ε, Ε, διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε μια συνολική αξιολόγηση των εποπτικών της ικανοτήτων. Η πλειονότητα των παραβιάσεων, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, σχετίζεται με το χρόνο εφαρμογής και μεταφοράς στο Εθνικό Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Και καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι οι γενικές διευθύνσεις ε, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες προκλήσεις. Γι' αυτό και χρειάζονται τη βοήθεια των κρατών μελών. Στους ελέγχους που θα διενεργούν χρειάζονται χρόνο. Η Κομισιόν δυστυχώς όμως δεν έχει ε, δώσει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγγελίες οι οποίες δεν τίθενται ποτέ σε επεξεργασία. Και όσον αφορά ε, ε, ε, την έναρξη διαδικασιών επί παραβάση. Δυστυχώ, πολλέ γενικέ διευθύνσει δεν έχουν απλώ τι γνώσει και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη προσδοκούν ότι θα χάνουν ε, ίση και δίκαιη μεταχείριση όσον αφορά την ε, παρακολούθηση τη ε, εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Γι' αυτό και ήταν μεγάλη μας χαρά που είχαμε στη διαδικασία αυτή τη δυνατότητα να συναντηθούμε με την ε, πρόεδρο της Επιτροπής σας αλλά και με την Ευρωπαϊκή... Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω άλλο, ούτε να σπαταλήσω το χρόνο σας. Όμως, θέλω να σας περιγράψω τι πιστεύω με ότι πρέπει να γίνει στο μέλλον από εδώ και πέρα. Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη, και αυτό αναγνωρίζεται και από την ίδια την Κομισιόν, η Κομισιόν να ενισχύσει περαιτέρω τις εποπτικές της δραστηριότητες σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συνθήκη. Και θεωρούμε ότι μπορεί η Κομισιόν να ενισχύσει και να προωθήσει και τις διαδικασίες απολογισμού που κάνει. Αυτό ε, επίσης βεβαίως ε, ακόμη και σήμερα ακούσαμε από την Κομισιόν ότι αναγνωρίζεται. Χρειάζεται περισσότερη συνέπεια, περισσότερο συντορισμό όσον αφορά την αξιοποίηση των ενωσιακών κονδυλίων η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μεταξύ των κρατών μελών είναι επίσης σημαντική. Το ίδιο και η κοινή χρήση των πόρων. Χρειάζεται συντονισμένη ροή πληροφοριών μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών όσον αφορά τις υποψίες ή και τις πραγματικές παραβιάσεις. Σίγουρα θετικό πάντως είναι το γεγονός ότι όλα τα κράτη-μέλη φαίνεται να είναι υπόλοιπα υπέρ της ε, περαιτέρω ανάπτυξης των εργαλείων προώθησης ευρωπαϊκής νομοθεσίας από πλευράς Κομισιόν. Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία σε αυτό. Η Κομισιόν βεβαίως θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με ε, την, τον χειρισμό από πλευράς της των υποθέσεων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερα σημαντική να, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση ανάμεσα στο δικαίωμα εμπιστευτικότητα ορισμένων πληροφοριών από πλευρά καρδομελών, αλλά και στη διαφάνεια αφετέρου. Έχουμε λοιπόν καταλήξει σε κάποιε παρατηρήσει, σε κάποιε σκέψει. Συνολικό πόρισμα όμως πρέπει να σας πω σε σχέση με τη μελέτη μας είναι ότι δεν πρόκειται για μια ε, εις βάθος ανάλυση όλων των διαστάσεων. Βεβαίω. Αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον και αυτό θα βοηθήσει στο να εντατικοποιήσουμε το έργο το δικό μας και το δικό σας. Εμείς δεν επιδιδόμαστε σε κυνήγι μαγισσών. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις συζητήσεις που έτσι και αλλιώς γίνονται σε διάφορα θεσμικά όργανα. Θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια χαρτογράφηση των βελτιστών πρακτικών σε επίπεδο κρατών μελών, κάτι που θα μπορούσε να ενδιαφέρει και εσά τους ευρωβουλευτέ. γιατί αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει συνολικά όλα τα θεσμικά όργανα και κυρίως τους πολίτες που είναι και το βασικό μας μέλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Ακούσατε και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις από τους ευρωβουλευτές εδώ. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η εφαρμογή, η θέση σε ισχύ του ενωσιακού δικαίου αποτελεί το θεμέλιο του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας σε όλα όσα είπατε. Είμαστε στο πλευρό σας. Εμείς σημειώσαμε όλα αυτά που παρουσιάζονται ε, στην ε, μελέτη σας. Θα διαβιβάσουμε τα πορίσματα αυτά και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και θέλω να σας διασφαλίσω ότι θα έχετε την αμέριστη στήριξη της Επιτροπής Αναφορών και στο μέλλον στις συζητήσεις που θα γίνουν. Ίσως θα πρέπει και στο μέλλον να δούμε αυτό το θέμα. Το θέμα της αποτελεσματικότητα της εφαρμογής από πλευράς κρατών μελών των αποφάσεων και των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Ε, αναφερθήκατε και σε μια πιθανή μελλοντική μελέτη σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλώς kollégák, Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα θέλω να προχωρήσουμε στη συζήτηση δύο συγκεκριμένων αναφορών. Η πρώτη είναι η 0228 του 2017, Παύλο Τούση είναι αναφέρον και αφορά την διατήρηση ε, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδα στην περιφέρεια της Λιγουρίας στην Ιταλία. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Τόση. Είναι παρόν. Γεια σας, σας καλωσορίζω κύριε Τόση. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους με αυτή την αναφορά. Θέλουμε να αναφέρουμε στα 20 και 227 της συνθήκης όσον αφορά την ε, παραβίαση του κοινωτικού δικαίου για την προστασία των ε, φυσικών και ή μη φυσικών βιοτόπων, οικοτόπων και την προστασία χλωρίδας και πανίδας αυτής της περιοχής. Και πολλές φορές ε, γίνεται η, αξιολόγηση των επιπτώσεων μόνο σε έργα που αφορούν την ε, περίμετρο των τοποθεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Εδώ έχουμε διάφορα προβλήματα. Έχουμε μια χωματερή στο Σαναρέμο, έχουμε επίσης την αποκατάσταση, αναμόρφωση του κόλπου του Σαν Μιγέλες Δωραπάλο, επίσης ε, τη βυθοκόρηση όσον αφορά τον κόλπο του Λεβάντο, του, της Μάγκρα και επίσης ε, του Παρόντι και Φόρνατζε. Και δεν αρκεί αυτή η παρέμβαση να αφορά ε, την Ποσειδονία ή μια τοποθεσία ενδιαφέροντος του Natura 2000 ούτως ώστε να ισχύει η υποχρέωση της αξιολόγησης επιπτώσεων. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, όπως λέει η νομοθεσία, να έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης επί της ουσίας για το έργο, σχέδιο, πρόγραμμα και να μην υπάρχει κάποιο είδους ε, ε, διαδικαστικού τυπικού χαρακτήρα ενέργεια όσον αφορά την προστασία της περιοχής όπου θα γίνει το κάθε φορά έργο. Οπότε τώρα έχουμε το οικόπεδο 6 του Σανρέμου που υπάρχει εκεί σχετική ε, χωματερή και εδώ επίσης έχουμε μια σπηλιά που έχει θεωρηθεί τόπος κοινωνικού ενδιαφέροντος και επίσης ε, έχουμε ε, την απόφαση 705 και 613 τις αποφάσεις που αφορούν ε, την κοιλάδα αρμία, το δηλαδή ένα κομμάτι αυτής. Βλέπετε εδώ μια φωτογραφία και πάμε τώρα στη θυμισμένη περιοχή Τσίνκουε Τέρε και εδώ λέμε ότι υπάρχει το κριτήριο του να μην υπάρχει εξολόγηση για τα 15 μέτρα και έχουμε την απόφαση 1459 ε, συγγνώμη εδώ πέρα γίνει ένα τυπογραφικό λάθος και λέμε ότι εδώ θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ενδεχομένες συνέπειες και ότι ε, υπάρχει καταστροφή ευαίσθητων οικοτόπων λόγω της βυθοκόρησης ακόμη επίσης και για το ότι έτσι παροξύνονται οι συνέπειες της ε, ε καταστροφής του, του, εδάφους. Ε, και ας μην συνδέεται αυτό άμεσα. Βλέπουμε τώρα την, τον κόλπο του Λεβάντο και επίσης βλέπουμε ότι έχουμε αυτές εδώ τις αεροφωτογραφίες που έχουν σχέση με ε, αυτό τον όρμο ε, αυτό το αυλάκι τέλος πάντων και ε, εδώ είναι μια διαφορετική ζώνη, ξεχωριστή από την ε, τοποθεσία κινητικού ενδιαφέροντος που είπαμε προηγουμένως. Παρακάτω έχουμε το αυλάκι φορνάτσε και δεν έχει γίνει και εκεί αξιολόγηση επιπτώσεων έχουν γίνει κινήσεις και έργα. Και αυτό παρά το ότι εκεί που όμορο σε αυτή την περιοχή υπάρχει μια τέτοια τοποθεσία κινητικού ενδιαφέροντος. Και εδώ, σύμφωνα με το ΙΟΤΑΤΑΒ 1345, έχουμε την σπηλιά της Αρκούδας που καλύπτεται από το εθνικό κτηματολόγιο. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά ε, βλέπετε τις φωτογραφίες από τη Λιγουρία. Τώρα για να δούμε εδώ τι γίνεται όσον αφορά αυτή τη βυθοκόρηση του τελευταίου κομματιού. Έχουμε ε, την απόφαση για το 34 που είναι η σχετική τοποθεσία κινητικού ενδιαφέροντος και τέλος έχουμε την αποκατάσταση αυτού του, του κόλπου Ραπάλο που αποτά επίσης προστατευόμενη περιοχή και εδώ έχει, έχει τα λεγόμενα λιβάδια της ε, ε, Ποσειδονίας ε, πάνω σε βραχώδες ε, υπέδαφος το οποίο είναι σημαντικού πάχους και όλα αυτά βλέπουμε ότι παρά την σε θέση με τόπο κοινωνικού διαφέροντος δεν έχουμε αξιολόγηση επιπτώσεων και σας ευχαριστώ Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Τόση. Ο Κελεάντικο είναι εδώ μαζί μας, ε, νομίζω, ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τον αναφέροντα που μας τα είπε όλα αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει τέτοια διαμαρτυρία ε, για το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Έχουμε ένα σωρό καταγγελίες ούτως ώστε το 2014 αρχίσαμε μια έρευνα και αφετηρία ήταν ακριβώς αυτές οι καταγγελίες τις οποίες και εξετάσαμε ε, βέβαια κάποιοι ισχυρισμοί ήταν αβάσιμοι αλλά κάποιοι άλλοι απεκάλυψαν και ανέδειξαν ένα πρόβλημα συγκεκριμένο που αφορά ε, περιφέρεια, που αφορά συγκεκριμένες τοποθεσίες. Οπότε γι' αυτό και ε, αρχίσαμε επαφές με την κυβέρνηση, ούτω ώστε να δούμε ε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές πώς θα εφαρμοστούν κατευθυντήριες που υπάρχουν και αυτό το άρθρο, το 6.3, για να μπορέσουμε να δούμε εις βάθος την κατάσταση αυτή που μόλις μας περιέγραψαν και συνέχισαν, συνεχίσαμε τις επαφές, ε, υπήρξαν παρατηρήσεις και πώς θα να δούμε αν μπορούμε να τα διασταυρώσουμε όλα αυτά και να έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν θα είμαι έτσι τυπολογικά να δούμε τα πράγματα τυπολατρικά, αυτό με τα 15 χιλιόμετρα και λοιπά. Θέλουμε να δούμε ακριβώς τι διαχείριση έγινε για την κατάσταση. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παράση, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα που ακριβώς όπως μας είπε η Επιτροπή είναι δύσκολο έγινε ολοσχερής αγνόηση εδώ της κοινωτικής νομοθεσίας όσον αφορά αυτές τις τοποθεσίες που θα έπρεπε να προστατεύονται σύμφωνα με το κοινωτικό δίκαιο. Πρόκειται για την ε, οδηγία των βιοτόπων οικοτόπων συγκεκριμένα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο το διαπιστώνουμε ότι συντρέχει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία και σε αυτή την περίπτωση στην Λιγουρία. και είναι σημαντικός ο αριθμός των περιπτώσεων που έχουμε παραβίαση ή απλώς μη εφαρμογή των κινητικών οδηγιών ή έχουμε στρεβλή εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους. Συγκεκριμένα δεν είχαμε αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα έργα, σχέδια αυτά που πρέπει να γίνεται όποτε έχουμε ε, τοποθεσίες κοινωτικού ενδιαφέροντος. Το αποτέλεσμα είναι σορευτικό από κάποιο έργο ή πρόγραμμα. Είναι από πολλές κατευθύνσεις και περισσότερες οι δραματικές συνέπειες ε, ενός ε, έργου στην ε, περιοχή, στη βιοπικιλότητα, στο νερό. Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει κάτι να γίνει μια που υπάρχουν τόσες ενδείξεις, τόσες ετήσιες εκθέσεις της περιβαλλοντικής υπηρεσίας Ένωση που δείχνουν ότι τα πράγματα επιδεινώνονται. Είναι σε κατάσταση, σε φάση κρίσης σε κάθε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό, παντού. Άρα θα πρέπει να γίνεται σωστή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της νομοθεσίας για τη φύση, για το περιβάλλον. Συζητήσαμε πριν με τους εκπροσώπους του ελεκτικού συνεδρίου ενδιαφέροντα πράγματα. Να, πώς σχετίζονται εκείνα με τη συγκεκριμένη οδηγία για την προστασία της φύσης για το Natura 2000 για τις περιοχές του κλπ. Και έχουμε αυτά τα 47 έργα τα οποία αξιολογούνται, αλλά από αυτά μόνο 7 από τα 47 είχαμε τη σωστή αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ε, πολύ λίγα. Βλέπετε τη διάσταση του προβλήματος που είναι πανευρωπαϊκό. Άρα θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά το κοινωτικό δίκαιο. Να λάβουν υπόψη τις σωρευτικές συνέπειες που, γίνονται, που υπάρχουν. Να προσπαθήσουν περισσότερο και οι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που μαθαίνω ότι υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα και θα δημοσιοποιηθούν σύντομα από πλευράς Επιτροπής. Άρα αυτό να δούμε. Τι γίνεται με την αποκατάσταση, την αναμόρφωση του και κλπ. Τι γίνεται από την αποκατάσταση από την τεράστια ζημία που έχει α, δημιουργηθεί εκεί στο περιβάλλον, στο έδαφος. Θα πρέπει να απευθυνθούν οι σωστές επιστολές προς τις περιφερειακές αρχές θα πρέπει να ζητηθεί η σωστή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Και μόλις όλα αυτά έχουν γίνει, μόλις έχουμε ε, αυτά τα έγγραφα προσανατολισμού, αυτό να κάνουμε κι εμείς. Να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Στο μέλλον να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί. Βέβαια, είναι και θέμα της διαδικασίας κατά της Ιταλίας για παράβαση του κοινωτικού δικαίου. Α, μισό λεπτό να το διορθώσω. Η διαδικασία EU Pilot αφορά το ότι δεν έγινε σεβαστή η νομοθεσία για το Natura 2000 και τις περιοχές που χρήζουν προστασίας. Είναι κληρονομιά αυτή που πρέπει να προστατεύεται. Άρα θα μείνει, να μείνει ανοιχτή αναφορά και να απευθυνθούμε όπως πρέπει σε αρμόδιες αρχές. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Όχι. Όχι, με συγχωρείτε. Ο κύριος Γιάρ. Πολύ σύντομα. Ε, στο, στα έγγραφά μου ε, είχα την αναφορά ότι θα μπορούσαμε να, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ίσως όμως μιλάμε για μια επιτυχημένη ιστορία. Η Κομισιόν αναγνωρίζει το πρόβλημα, συντάσσει και κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ που δεν, είναι, δεν έχουν οριστικοποιηθεί πλήρω, αλλά βρίσκονται στο τελικό στάδιο τη επεξεργασία του. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να την κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ξαναδούμε το θέμα όταν οριστικοποιηθούν αυτέ οι κατευθυντήριες γραμμέ. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτέ οι κατευθυντήριες γραμμές θα κατατείνουν προ την εξειδίκευση και την ερμηνεία ε, τη ε, νομοθεσία, Νομίζω Ορθώς είπε η Κομισιόν ότι δεν ε, συνοδεύεται κάθε καταγγελία από πραγματική διαπίστωση παραβίασης. Όμως αναγνωρίζει η Κομισιόν ότι χρειάζεται ενδεχομένως να δοθεί μια πίεση, να, να δοθεί μια όθηση αν θέλετε. Γι' αυτό και συντάσσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Προφανώς μπορούμε να παραμείνουμε και σε επαφή με τον ε, αναφέροντα ώστε να μας ενημερώσει σχετικά με το αν ο ίδιος διαπιστώσει κάποια πρόοδο, κάποια βελτίωση σε σχέση με τα πράγματα, άπαξ και εκδοθούν και αρχίσουν να εφαρμόζονται συγκεκριμένε κατευθύνες γραμμές. Οπότε ας μείνει ανοιχτή. Κύριε Τόση, σας ξαναδίνουμε το λόγο για να μας απαντήσετε. Χίλια ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό αυτό το οποίο άκουσα από τους ε, βουλευτές μέλη της Επιτροπής σας και θεωρώ ότι ε, το Προεδρείο της Επιτροπής θέλει να μην ανοιχτεί η αναφορά θέλει να αφήσει την πόρτα ανοιχτή και καθώς μια φορά θεωρώ ότι αυτό είναι χρήσιμο είναι δίκαιο και είπαμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας ε, τους ε, μέλλοντες ε, κανόνες που θα διέπουν το πρόβλημα το οποίο αφορά η αναφορά μου. Είμαι από την Λιγουρία και ακριβώς εκεί κατοικώ. Εκεί σε αυτές τις περιοχές που αφορά η σημερινή αναφορά. Οπότε θα μπορούσα και στο μέλλον να συμβάλλω τόσο ώστε να τηρηθούν οι δέουσες διατάξεις. Και σε αυτό να συμβάλλουν όλοι οι συναρμόδιες αρχές. Ευχαριστώ και πάλι. Ωραία, σας ευχαριστούμε κύριε Τόση. Και εγώ κρατώ ως θετικό τη στάση της Κομισιόν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη μου τα σχόλια των συναδέλφων, κρατάμε ανοιχτή την αναφορά, θα αποστείλουμε επιστολή στις Ιταλικέ Αρχές, θα τους θέσουμε το θέμα, θα συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίε, θα απευθυνθούμε και στις, ε, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και στις τοπικές αρχές της Λιγουρίας, θα τους θέσουμε αυτό το θέμα, θα παρακολουθήσουμε ποιες, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχει αυτός ο διάλογος ε, στην πράξη και αν οι εμπειρογνώμονές μας καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα και να το ξαναδούμε, ε, θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας, ε, να σας ικανοποιεί και σας κύριε, αυτή η στάση. Η Τσέντε πότε θα πάμε στην επόμενη αναφορά. 0754. Ισπανικής Ιθαγένειας και το θέμα της αναφοράς αυτής είναι η απόρριψη ανεπεξέργαστων λιμάτων στο φυσικό πάρκο Λαμαριάλ Πεγκολίβα. Θέλω, κύριε Αλεμανή, ε, καταρχάς να ρωτήσω, είστε εδώ? Α, ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο λοιπόν. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας. Μας δίνετε ευκαιρία να το πετούμε. Ονομάζομαι, όπως σωστά είπατε, Βιθέντε Πόρτες Αλεμάνη και ε, εκπροσωπούμε το προ Μοντεπέγο που είναι με ένας φορέας ε, της περιοχής του Αλικάντε. Έχουμε πάνω από 40 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, αυτή, αυτό, το οικοδομικό συγκρότημα, αλλά δεν έγινε αυτό που πρέπει να γίνει. Και έχουν εγκαταλειφθεί τελείως οι δημόσιες, οι ε, δημοτικές υπηρεσίες. Και όπως πέρασε ο χρόνος, τα πράγματα χειροτερεύουν όσον αφορά τις βασικότερες υποδομές. Ε, και πρόκειται για αυτό το, το χώρο καθάρισης των λιμάτων και των ε, υδάτων και κάθε μέρα έχουμε ένα σωρό μολυσματικά, ε, ρηπαντικά στοιχεία τα οποία πέφτουν εκεί σε αυτή την περιοχή που προστατεύεται από το Natura 2000. Κανένας, καμία αρχή δεν μπόρεσε να βρει και να δώσει κάποια λύση τόσα χρόνια. Παρά το ότι τόσα χρόνια έχουμε ενημερώσει τις τοπικές αρχές, τις αρχές της περιφερικής διοίκησης και τις κρατικές για το ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ε, λύματα, αυτά τα απορρίμματα. Ε, οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση που ε, να, να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση που είναι συνεχής. Άρα χρειάζεται άμεσα ε, ανάληψη δράσης και απευθυνθήκαμε ε, στην την κυρία περιφέρεια της ε, Βαλένθια και στις αρχές του αυτού του <clears throat> φυσικού πάρκου να αναλύσουν το pH, την θερμοκρασία, τη χλωροφύλλη, το περιεχόμενο σε άλλας, σε άλατα τέλος πάντων σε μία ζώνη δύο χιλιόμετρων από εκεί που πέφτουν όλα αυτά τα σκουπίδια και να δούμε κατά πόσον έχουμε ρήπανση και μόλυνση του φυσικού πάρκου. Ε, τελικά έδειξε η ανάλυση ότι αυτό είναι αλήθεια, ότι, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, γιατί 43 φορές περισσότερο από ότι πρέπει τα, ε, ε υπάρχουν αυτά τα e-coli και 72 φορές περισσότερα ε, ε ακάθαρτα στοιχεία. 1.500 Τα υλικοβακτηρίδια και άλλα βακτηρίδια τέλο πάντων μολυσματικά και είπαμε ότι όλα αυτά φύγουν την ε, οικιστική ζώνη του Μοντεπέγο όπου υπάρχουν πάνω από 1.500 ε, κατοικίες οπότε έτσι έχουμε παραβίαση της ε, οδηγίας για τα πτηνά, για τα, τους οικοτόπους, για τα ύδατα και τώρα υπάρχει η περίπτωση να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ζημία όσον αφορά ε, τις οριζοκαλλιέργειες ή όσον αφορά το πόσιμο νερό που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά εκεί στην περιοχή Ντένια. Ε, ελπίζουμε ότι σημερινή μας επίσκεψη θα είναι το ποσιμο νερο που βρισκονται παρα πολυ κοντα εκει στην περιοχη ντενια βήμα για να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Αλεμάνι, Κύριε Φλωρίδο, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτή την αναφορά καταγγέλλεται το ότι κατευθύνουν ακάθαρτα νερά εκεί στην επαρχία του Αλικάντε στη διοικητική περιφέρεια της Βαλένθια όπως είπε ο αναφέρον. Τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε εξετάσει την αναφορά πώς μας την διαβιβάσατε. Λάβουμε υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης που συντρέχει όσο αφορά το δίκαιο και είπαμε όσον αφορά ε, την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και των υδάτων. 91 του 271 είναι σχετική οδηγία για τα λίμματα και ακριβώς εδώ έχουμε αυτό το, το, το, την αστική περιοχή, το οικοδομικό συγκρότημα ε, είναι τα κριτήρια, το, το μέγεθός τους για να δει κανείς αν συντρέχει εφαρμογή της οδηγίας. Οπότε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε που μας διαβίβασε η Ισπανία, αυτή η οικιστική περιοχή, το Μοντεπέγο, από όπου προέρχονται αυτά τα, τα κάθαρτα ε, υλικά δεν έχει χαρακτήρα ε, αστικής περιοχής γιατί έχει κάτω από 2.000 κατοίκους και η οδηγία άρα δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει επίσης ο Δήμος του Πέγο, εκεί υπάγεται. Ο Δήμος του Πέγο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα τηρεί τα όσα επιτάσσει η οδηγία. Σας επισημαίνουμε ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τι κάνουν τα κράτη-μέλη και αν εφαρμόζουν αυτή την σημαντική οδηγία για προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ακριβώς αναφέρθηκε αφορά και την υγεία, την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων αλλά και οικονομική δραστηριότητα όπως τουρισμός και γεωργία για την Ισπανία συγκεκριμένα έχουμε τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια βελτίωση, αλλά έχουμε και στραβοπατήματα στην, στην εφαρμογή της οδηγίας. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ξεκινήσει κάποιες οριζόντιες διαδικασίες παραβάσεων που αφορούν πολλές ε, αστικές περιοχές στην Ισπανία και γίνει προσφυγή ε, κατά της Ισπανίας ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Α, τώρα το καλογέρι υπευλήθησαν οι οικονομικές κυρώσεις στην Ισπανία κατόπιν σχετική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου. Τώρα πάντως για τον Δήμο του Πέγο δεν ε, έχουμε περίπτωση εφαρμογή του σχετικού κοινοτικού δικαίου. Τώρα όσον αφορά την προστασία, ε, έχουμε εδώ το Μαργάλ Πεγολίβα ε, που υπάρχει στο Natura 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεκήρυξε αυτό, αυτή την περιοχή ως μέλος, μέρος α, του, προστα... του δικτύου που θα πρέπει να προστατευτεί γιατί αφορά το φυσικό περιβάλλον και έχουμε εδώ κάποιους φυσικούς πόρους, υπάρχει νομοθεσία του 2004, έχουμε κανόνες, έχουμε υποχρεώσεις, όπως το ότι λίμματα έργα δεν θα πρέπει να κατευθύνονται προς τα εκεί και ότι θα πρέπει να υπάρχει προστασία και των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή. Επομένω, συμπερασματικά, επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαπιστώνει παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Δεν υπάρχουν στοιχεία να θεωρήσουμε ότι έχει υπάρξει κάτι που αποτελεί κακοδιαχείριση του φυσικού πάρκου. Επίσης, πρόσφατα επέβαλαν κυρώσεις οι Ισπανικές αρχές για τέτοιου είδους ε, ακάθαρτα στοιχεία τα οποία ε, εκβράζονται, τα οποία ε, προωθούνται προς το πέγο. Βλέπουμε επομένω ότι αυτές οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά για να ισχύσουν το κοινωτικό δίκαιο να αποδίδουν οι καταγγελίες που γίνονται και όποτε χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει στο δικαστήριο αλλά στις καταγγελίες που έχουμε κάνει και προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, δεν περιέχει, δεν καλύπτεται ο Δήμος του Πέγου. Ευχαριστούμε πολύ για την περιγραφή της κατάστασης. Ο κύριος Τερικάμπρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Τερικάμπρας. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο θέλει ο αναφέρον, αλλά είναι ξεκάθαρη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρη στην ασάφειά της. Άρα πρέπει να κάνουμε και να προβληματιστούμε. Είναι σαφές λοιπόν ότι καταρχήν το Ισπανικό κράτος δεν έχει σωστή διαχείριση καθαρισμού των υδάτων. Είναι χίλιες οι περιπτώσεις ε, των, μαύρων ζωνών των επιλείψιμων σημείων στην Ισπανία σχετικά με αυτό. Μα τι γίνεται. Το, κριτήριο μας βλέπετε του Πέγο είναι το αν ε, αυτή η περιοχή, το Πέγο μάλλον η περιοχή προκαλεί το, πρόγραμμα, το πρόβλημα ε, υπάγεται στο πέγο ή αν είναι διοικητικά, οικιστικά, ανεξάρτητη. Και έτσι θα κρυφθεί το αν θα υπάρχουν κυρώσει για το αν θα εφαρμοστούν. Μα δεν ξέρουμε τι έχει εφαρμοστεί. Να, η ασάφεια. Οπότε λέτε ότι ο Δήμος καταλήγεται κάνει ό,τι πρέπει. Περίεργο. Μα αφού έχουν ήδη επιβληθεί ε, κυρώσεις από το κράτος για παραβάσεις. Άρα πώς δεν έχουμε παρανομία. Τώρα για την οικιστική αυτή, την αστική αυτή περιοχή έχει το κριτήριο αυτό των 2.000 κατοίκων. Ναι και αν έχουμε 1.500, τι γίνεται, 1.500 μάλλον ε, κατοικίες. Πώς έχουμε 1.500 σπίτια και 2.000 ε, ε, κατοίκους, 1,5 σε κάθε σπίτι. Δεν είναι δυνατόν. Και Μα ε, λίγο είναι και αυτό που συμβαίνει. Και αυτοί δηλαδή που υποφέρουν λίγοι είναι. Επίσης βρισκόμαστε κοντά σε ένα φυσικό πάρκο. Η Ένωση το προστατεύει. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε και από ό,τι φαίνεται αυτά τα λίμματα έχουν φτάσει στα 350 μέτρα από το φυσικό πάρκο και προχωράνε. Ε, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από όσα ξέρω αν είναι κάτι που κάνει είναι ότι προστατεύει το περιβάλλον. Ε, άρα θα πρέπει, θα πρέπει να προσέχουμε πολύ την υπόθεση περιβάλλον. Και προσωπικά θεωρώ ότι κάποιες οδηγίες έχουν παραβιαστεί και αφορούν την οργάνωση αυτής της υπόθεσης στο πέγο. Τα τοξικά στοιχεία, τα ρηπαντικά, μολυσματικά στοιχεία και άρα θα πρέπει πρώτα πρώτα μην είναι η αναφορά δεύτερον θα πρέπει να ξεκαθαριστούν ε, αυτά τα ασαφή σημεία θα πρέπει να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για ένα χωριό, μιλάμε μια ολόκληρη οικιστική ζώνη, οικοδομικό συγκρότημα, τι είναι. Πρόκειται για κάποιες παραβιάσεις που έγιναν. Το θέμα είναι αν ελήφθη δράση κατά αυτών των παρανομιών γιατί ζητήθηκε, ζητήθηκε να υπάρξει αντίδραση. Εάν δεν έχουν ξεκαθαριστεί όλα αυτά τα σημεία τότε έχει δίκιο ο αναφέρον να μας ζητεί την βοήθεια. Ε, εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Πρόεδρος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο. Ο κύριος Πέτερ πάνω που νόμιζα ότι είχα καταλάβει την απάντηση τη Κομισιόν, διαπιστώνω ότι δεν κατάλαβα. Εσείς είπατε τώρα ότι δεν υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκών οδηγιών, μεταξύ άλλων διότι εδώ πρόκειται για έναν πολύ μικρό οικισμό. Από την άλλη πλευρά η Κομισιόν είπε ότι περιμένει να, να αναλυφθεί δράση από την ίδια ή από τις Ισπανικές Αρχές. Ε, κάπως αυτά μάλλον δεν, δεν συνάδουν το ένα με το άλλο. Ε, ακούω και τους Ισπανούς συναδέλφους και σχηματίζω την εικόνα ότι σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, ακόμη και αν τελικά αυτό το πρόβλημα δεν εμπίπτει η επίλυσή του στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τις Ισπανικές Αρχές, να λάβουμε κάποιες πληροφορίες. Ίσως αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ίσως αυτό το, αυτό το, το, το μπέρδεμα στο μυαλό μου που μου προκάλεσε η Κομισιόν μπορεί να, να μου το διευκρινίσει. Αφενός δηλαδή δεν υπάρχει παραβίαση ε, κατεξοχήν της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από την άλλη όμως θεωρεί και η Κομισιόν ότι ε, ε, πρέπει να αναλυφθεί κάποια δράση. Δεν κατάλαβα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα την ε, εξής λύση. συνάδελφοι, κύριε Αλεμάνη, θέλω να σας πω το εξής. Πρώτον, υπάρχει πρόβλημα. Το αναγνωρίζουν οι πάντες. Υπάρχει πρόβλημα, το είπε και ο αναφέρον, το ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το θεωρεί δεδομένο ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αφού υπάρχει πρόβλημα, γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούμε να την κλείσουμε την αναφορά. Άρα, την κρατάμε ανοιχτή. Τρίτον, υπάρχουν μια σειρά από ανοιχτά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το αναγνώρισε αυτό και η Κομισιόν. Πρότασή μου λοιπόν θα ήταν να αποστείλουμε επιστολή στις Ισπανικές αρχές μέσω της οποίας θα ζητούμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Άπαξ και τις λάβουμε αυτές τις απαντήσεις θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε το θέμα και να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Διότι το να παίξουμε τώρα την κολοκυθιά με το τι είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, τι εμπίπτει, τι δεν εμπίπτει σε αυτήν, νομίζω ότι δεν είναι δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Ας ε, απευθυνθούμε λοιπόν σε μια πρώτη φάση στι ισπανικέ Αρχές και από εκεί και πέρα θα το ξαναδούμε το θέμα για το πώ θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ συνάδελφοι και περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης που είναι το σημείο 9. Έχουμε ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μαριά σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια θα ακολουθήσει συζήτηση, αλλά πρώτα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαριά. Ε, πραγματικά η γνωμοδότηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εξετάζει το πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνθήκης που αφορούν την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω, όταν πρόκειται για μια γνωμοδότηση επειδή υπάρχει και περιορισμένος όγκο στο τι μπορούμε να γράψουμε υποχρεωτικά έχουμε αναδείξει πέντε σημαντικά σημεία και φυσικά αναμένουμε τις τροπολογίες των συναδέλφων προκειμένου να εμπλουτιστεί η έκθεση. Αλλά η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική ιδίως στο σημείο 1 που αναφερόμαστε στα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε λίγους μήνες έχουμε και τις ευρωεκλογές. Επομένως δεν μιλούμε γενικώς θεωρητικά, αλλά μιλούμε πολύ πρακτικά. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι έχουμε μια περίπλοκη εκλογική νομοθεσία. Διότι η νομοθεσία για τις ευρωεκλογές είναι μεν προσδιορισμένη με απόφαση του ε, Συμβουλίου το 1975, αλλά κάθε κράτος μέλος προσθέτει ιδιαίτερες διατάξεις για την χώρα του. Οι διατάξεις αυτές όμως θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είναι αυθαίρετες. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση που κάνουμε είναι ότι πρέπει η νομοθεσία της ίδιας της ε, ε, των κρατών μελών για τις ευρωεκλογές τουλάχιστον να εγκρίνεται ένα χρόνο πριν τις ευρωεκλογές για να ξέρουν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες πώς θα συμμετάσχουν και με ποιους όρους. Δηλαδή το να αλλάζει ξαφνικά η νομοθεσία των ευρωεκλογών δύο-τρει μήνε πριν τι ευρωεκλογέ, επειδή σε κάποιο κράτο η κυβέρνηση βλέπει το συσχετισμό δύναμη και με βάση το συσχετισμό δύναμη αλλάζει την εκλογική νομοθεσία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι σοβαρό και δεν πρέπει να συμβαίνει. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι αν πρέπει να υπάρχει όριο εισόδου στις ευρωεκλογές. Δηλαδή πολλές χώρες έχουν ένα ποσοστό 3 ή 5% προκειμένου να μπορεί κάποια πολιτική δύναμη να εκλεγεί. Το ποσοστό εισόδου εφαρμόζεται σε εκλογικά συστήματα κυρίως όταν πρόκειται να δημιουργηθούν σταθερές κυβερνήσεις και για να έχουμε μια σταθερή πλειοψηφία στα εθνικά κοινοβούλια. Εδώ όμως στην Ευρωβουλή δεν έχουμε τέτοιο σύστημα, άρα η δημιουργία ενός threshold 3%, 5% επί του πρακτέου αφαιρεί το δικαίωμα από τους πολίτες να μπορούν να εκφραστούν πλήρως και κυρίως από τις μικρές σε δύναμη πολιτικές ομάδες να μπορούν να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογέ. Έτσι λοιπόν το θεωρώ αυτό το σημείο ως απαγορευτικό και έμεσο τρόπο αποκλεισμού όλων των απόψεων που δεν είναι πλειοψηφικές. Το δεύτερο ερώτημα είναι τα συμβίβαστα που υπάρχουν ή τα κολλήματα. Εγώ είμαι από την Ελλάδα, ο συνάδελφός μου δίπλα είναι, που θα μιλήσει για το SND είναι από την Κύπρο. Στην Ελλάδα, προκειμένου να είσαι υποψήφιος στις ευρωεκλογέ, εάν είσαι βουλευτής, όπως ήμουν εγώ το 2014 πρέπει να παρετηθείς πρώτα από βουλευτής και εν συνεχεία να έχει το δικαίωμα να είσαι υποψήφιος. Αυτό ισχύει μόνο στην Ελλάδα και στη Λετωνία. Αντίθετα στην Κύπρο κάποιο που είναι βουλευτής μπορεί να είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτή και αν εκλεγεί να διαλέξει τι από τα δύο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμά στην Ελλάδα μας περιορίζει τα δικαιώματα. Και εγώ παρετήθηκα από εθνικός βουλευτής το 2014 απλά για να είμαι υποψήφιος. Θα μπορούσα να μην είχα εκλεγεί, οπότε έτσι θα είχα παρετηθεί και από βουλευτής και από ευρωβουλευτής. Το άλλο θέμα που υπάρχει είναι αν πρέπει να έχουμε λίστα ή σταυρό προτίμηση. Διότι όταν υπάρχει λίστα, και σε πολλέ χώρε υπάρχει λίστα, η απόσταση ανάμεσα στου πολίτε και στου εκλογεί και στου βουλευτές είναι μεγάλη. Διότι στην ουσία σε κλειστά ε, δωμάτια οι κομματικές ηγεσίε επιλέγουν τη λίστα χωρίς να έχουν την ευκαιρία οι πολίτε να επιλέγουν με σταυρό προτίμησης. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα και σε μερικές άλλες χώρες έχουμε σταυρό προτίμησης. Αυτό το θεωρώ κατάκτηση, αλλά βλέπω ότι η ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια να καταργήσει το σταυρό προτίμησης και να επαναφέρει τη λίστα. Ίσως γιατί αρκετοί ευρωβουλευτές είναι ενοχλητικοί προ τι ηγεσίε του. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί, γιατί δεν μπορεί να αλλάζει τους όρου του παιχνιδιού πέντε μήνες, έξι μήνες πριν τις ευρωεκλογέ, είναι ότι ετοιμάζουν σενάρια στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να κόψουν την χώρα σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες. Ενώ η Ελλάδα είναι μία εκλογική περιφέρεια για 21 ευρωβουλευτές, τώρα αρχίζουν σενάρια να δημιουργήσουν ένα κομμάτι για τη Βόρεια Ελλάδα, ένα κομμάτι για τη Νότια Ελλάδα και όλα αυτά γιατί. Για να μην μπορούν να εκφραστούν οι μικρές πολιτικές δυνάμεις. Γιατί αν κάποιες πολιτικές δυνάμεις πάρουν τουλάχιστον το 3%, όταν κόψει σε 2, 3, 4 εκλογικές περιφέρειες, τότε αυτοί δεν θα μπορέσουν να εκλεγούν. Εδώ λοιπόν έχουμε μία παρατήρηση ότι πρέπει να σταματήσουν αυτά τα τρίκ. Και αυτά τα τρίκ θα σταματήσουν αν υποχρεούνται οι κυβερνήσεις να μην αλλάζουν τον εκλογικό νόμο παρά ένα έτος πριν τις ευρωεκλογές. Σε μερικές χώρες αυτό υπάρχει. Σε άλλες όμως γίνεται μία, αν θέλετε, καιροσκοπική λειτουργία. Το επόμενο θέμα που αφορά το εκλέγεν και εκλέγεστε είναι ποιοι ψηφίζουν. Ποιο είναι το εκλογικό σώμα. Είναι δυνατόν ξαφνικά να μετατραπούν, να μετατραπεί το εκλογικό σώμα, δηλαδή να δοθεί δυνατότητα ας πούμε σε πρόσφυγες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μια χώρα ή σε κάποιους άλλους να αποκτήσουν την εθνική ηθαγένεια και έτσι να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογέ. Διότι σύμφωνα με τη συνθήκη το ποιος παίρνει την εθνική ηθαγένεια είναι αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Αλλά όταν ξαφνικά την εθνική ηθαγένεια ας πούμε στην Ελλάδα την πάρουν 800.000 άτομα με ελληνοποιήσεις που θα γίνουν Αλβανών, Πακιστανών και προσφύγων τότε δεν έχει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει. Δεν αλλάζει το εκλογικό σώμα. Δεν αποκτούν αυτοί δικαιώματα ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και European citizenship. Αυτό δεν αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Τίμερμανς, γιατί το έθεσε αυτό το θέμα, είπε ότι αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν δεν μπορείς ξαφνικά να ανοίγει τον κατάλογο των εκλογέων όποτε σου αρέσει και όπως σου αρέσει. Όπως επίσης έχουμε το αντίθετο. Κάποιες χώρες αποκλείουν ορισμένους πολίτες που δεν ζουν στη χώρα τους από το να ψηφίζουν. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη πριν 10 μέρες στο Στρασβούργο, όπου είδαμε Φερρυπίν στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες όσοι δεν κατοικούν στη συγκεκριμένη χώρα δεν μπορούν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογέ. Ούτε αυτό είναι σωστό. Εγώ νομίζω ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο θα πρέπει να μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Παραδείγματο χάρη η Ελλάδα λέει για τους πολίτες, τους Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι, ας πούμε, στο Βέλγιο, ότι μπορούν, αν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ελλάδος, εδώ στο Βέλγιο να πάνε στην πρεσβεία της Ελλάδος, στις Βρυξέλλες και να ψηφίσουν κατά τις ευρωεκλογές. Με ελληνικό ψηφοδελτίο. Ή οι Έλληνες πολίτες μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του Βελγίου και να ψηφίσουν πάλι στις ευρωεκλογέ, αλλά θα ψηφίσουν βελγικό ψηφοδέλτιο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλο και περισσότερους πολίτες της Ένωσης να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογέ. Και εδώ υπάρχει και η σκέψη Φερρυπίν για τους Έλληνες ομογενείς που κατοικούν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Καναδά, στην Αυστραλία, αν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να μπορούν στην πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον ή στο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη να ψηφίσουν. Το ίδιο και για την Αυστραλία. Αυτά όλα τα δικαιώματα και φέρνω παράδειγμα την Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι ισχύει για πολλέ χώρε. Για να μπορούμε να επεκτείνουμε τα δικαιώματα. Διότι ο στόχο είναι το δικαίωμα του εκλέγην να είναι απρόσκοπτο, το δικαίωμα του εκλέγεστε να είναι απρόσκοπτο, το εκλογικό σώμα να αναπτύσσεται με βάση το ποιοι είναι οι πολίτες του κράτους μέλους, αλλά όχι με τρίκ ελληνοποιήσεων και παρανόμων αν θέλετε διαδικασιών χορήγησης ηθαγένειας και το άλλο είναι ποιος προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί αναφέρουμε εδώ στο σημείο 1 ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει και να προωθήσουμε την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, δεν έχει καμιά αξία τι κάνουμε εμείς εδώ αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν το προβάλλουν εάν δεν εξηγούν τις απόψεις μας. Εάν όταν πάμε πίσω στη χώρα μας, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, δεν μας δίνουν το δικαίωμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκφραστούμε. Εάν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν μόνο συγκεκριμένα κόμματα και εξαφανίζουν όλους τους άλλους. Εδώ τι θα γίνει. Αυτό το θέμα της πολυφωνίας το έχω θέσει πάρα πολλές φορές σε αυτήν εδώ την αίθουσα την προηγούμενη εβδομάδα στη δημόσια ακρόαση είχαμε τον πρόεδρο της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ελληνικής και του επεσήμανα ότι όσον αφορά το ECR που είμαστε 10% της δύναμης δεν προβαλόμαστε ανάλογα από τα μέσα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε άλλα κράτη που δεν τους προβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο τι θα κάνει. Θα καθόμαστε να κοιτάμε και τι θα γίνει. 20 μέρες πριν τι εκλογές θα μας πούνε βεβαίως όλοι θα προβάλλεστε. Ναι, αλλά τέσσερα χρόνια μας έχουν εξαφανίσει. Πώ θα γνωρίζει ο πολίτη ποια είναι η δραστηριότητά μα, πώ θα γνωρίζει ποιε είναι οι πολιτικέ θέσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι και με γιατί η εισήγηση αυτή ήταν σύντομη, με πρέπει να διασφαλίσουμε το δικαίωμα τη πολυφωνία, το δικαίωμα του πλουραλισμού, το δικαίωμα να ακούγονται όλε οι απόψει. Αλλιώ είναι κοροϊδία οι ευρωεκλογέ. Αν δηλαδή δεν μα επιτρέπεται να ασκούμε τα δικαιώματά μας ως εκλογής αν αλλάζουν με τρίκ τον εκλογικό νόμο, αν δεν μας επιτρέπουν μέσα στα μαζικά μέσα ενημέρωση να ακουγόμαστε, τότε τι εκλογέ είναι αυτέ. Πρόκειται για εκλογέ φάρσα. Λοιπόν, γι' αυτό Θέλω να είμαι πολύ πρακτικός, θα έχω και τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα που έχει η έκθεση. Φυσικά η έκθεση αυτή αναφέρεται και στη δυνατότητα της εκλογικής εκστρατείας, στο σημείο 2. Στο σημείο 3 αναφερόμαστε στο δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε στις δημοτικές και τοπικές εκλογές, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό δικαίωμα, δηλαδή ένας ε, Ιταλός πολίτης να μπορεί να είναι υποψήφιος για εκλογικό αξίωμα Δήμου εδώ στο Βέλγιο, λέω παραδείγματο χάρη. Το επόμενο σημείο 4 είναι η δράση της Επιτροπής Αναφορών, την οποία όλοι γνωρίζουμε, σε σημαντικά θέματα όπως είναι τα θέματα, τα δικαιώματα του παιδιού, η απασχόληση, η ελεύθερη κυκλοφορία και τέλος, και κλείνω με αυτό, το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί. Έμεινα στο πρώτο σημείο διότι σε λίγους μήνες έχουμε ευρωεκλογέ. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα fake news που είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις, απόψεις μας, όταν εξαφανίζουν τη δραστηριότητά μας εδώ. Πώ θα κρίνουν οι πολίτε. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά θέματα. Αναμένω τις γνώμε και τις απόψεις των συναδέλφων για να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη έκθεση, η οποία νομίζω ότι όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε για τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να τοποθετηθώ ως σκιώδης, όχι ως ε, προεδρεύων του ΕΛΚ. Κύριε Μαριά, καταρχάς εκτιμώ βαθύτατα ε, τις εκκλήσεις που κάνατε. Νομίζω ότι περιγράψατε εξαιρετικά τα προβλήματα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις σας διαβεβαιώ ότι το ΕΛΚ συμφωνεί με αυτά που είπατε. Βεβαίως θα το συζητήσουμε και εσωτερικά στην πολιτική μου ομάδα και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε και σε μια συγκεκριμένη θέση ή σε ένα σύνολο θέσεων. Νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να γεφυρώσουμε τη θεωρία με την πράξη. Να εξασφαλιστεί η συνένεση και συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει μια σκηνή προσέγγιση απέναντι σε αυτές τις προσδοκίες και απαιτήσει που και εσεί περιγράψατε, κύριε Μαριά. Ε, τις επόμενες ε, εβδομάδες μάλιστα θα τοποθετηθούμε και γραπτός επί των θεμάτων αυτών. Θα ξεστήσουμε τα θέματα αυτά και στην, ε, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Θα υπάρχει και η σχετική ψηφοφορία της, για τη γνωμοδότησή σας το, στις 21 Νοεμβρίου. κύριος Παπαδάκης, εκ μέρους των Σοσιαλιστών, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Νόδη Μαριά, για το συνεχτικό κείμενο που <coughs> ετοίμασε. <coughs> Με συγχωρείτε. The next one later. Ο κύριος Παπαδάκη θα πάρει το λόγο στη συνέχεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ίσως ένα ποτηράκι ούζο, λέει ο πρόεδρος. Θα βοηθούσε. Τελικά άντε εγώ μέχρι να αναρρώσει. Συμφωνώ, συμφωνώ με τα περισσότερα που είπε ο κύριος Μαριάς. Όχι βέβαια να μην υπάρχει αλλαγή του εκλογικού δικαίου. Θα πρέπει να ισχύσουν τα παλαιά. Δεύτερον, τα εμπόδια για τους υποψηφίους ή ε, θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία για τα κολλήματα. Γιατί υπάρχουν υποψήφοι που έχουν πλεονέκτημα γιατί πατάνε σε δύο βάρκες. Τώρα όσον αφορά τους φραγμούς τα κολλήματα, ποιος καταρτίζει τη λίστα των κολλημάτων, πάντως το κατόφλι. Το κατόφλι είναι ένα ναυάγιο, μια τραγωδία, διότι θα αφήσει απ' έξω εκατομμύρια ψηφοφόρων. Ευτυχώς δεν θα ισχύσει για αυτές τις εκλογές του 19. Όμως, όμως, η κρίσιμη λέξη που ανέφερε ο Μαριάς ήταν η λέξη συμμετοχή και θεωρώ ότι αφού μας λέει κάτι για τους πολίτες εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε πολίτες συνεχώς, όχι μόνο όταν έχει εκλογές και ψηφίζουμε ούτε τα δέκα τρόλτα που παίρνει να ρίξει την ψήφο στην κάλπη Άρα, αν δεν αρχίσουμε να είμαστε πολίτες, στο τέλος δεν θα είμαστε ποτέ πολίτες. Αυτό θα είναι τραγωδία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κανείς ενεργός πολίτης στην Ευρώπη, να συμμετέχει, μην υπάρχει αυτό το όριο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει, θα πρέπει αυτό να τονιστεί στο τελικό κείμενο. Α, μισό λεπτό. Κάτι λίγο διαφορετικό, αλλά όχι και τόσο, Πρόεδρε. Στο κείμενο του προηγουμένου αναφέροντος δεν του δώσαμε την ευκαιρία να δευτερολογήσει, να απαντήσει τέλο πάντων όπως πάντα κάνουμε ο αναφέρον δεν απάντησε όπως πάντα. Συνήθως έχει δύο λεφτάκια για να απαντήσει. Δεν του δώσαμε την ευκαιρία. Το σωστό θα ήταν όταν τελειώσουμε με αυτό το θέμα να του δώσουμε ευκαιρία να απαντήσει. Τον συντάκτη νομοδότηση τον κύριο Μαριά για το κείμενο αλλά και για το ότι αναφέρθηκε σε διάφορες παραδοξότητες όπου υπάρχουν στην Ελλάδα και μάλιστα προσβάλλουν να θέλετε και την ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, καλό είναι όλα αυτά να τα λέμε στον κατάλληλο χρόνο ούτω ώστε να δείχνουμε ότι αυτό το οικοδόμημα ακούει και σέβεται όχι μόνο σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Συμφωνώ για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης, καθώς και για την ανάγκη να καταστεί η εκλογική διαδικασία πιο προσβάσιμη και διαφανής για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να είναι πιο ξεκάθαρα τα όρια της Ένωσης και των κρατών μελών σχετικά με το δικαίωμα της αναφοράς. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να έχει πιο προσβάσιμες διαδικασίες για κάθε πολίτη. Το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει περισσότερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, όπως αναφέρεται στις συνθήκε, όπου οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με άξονα τους πολίτες και την πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση τους σε αυτές. Επίσης το Συμβούλιο θα έπρεπε να συνεδριάζει δημοσίως κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί του νομοθετικού σχεδίου. Είναι σημαντικό οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που από τη συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως του δικαιώματος τους στην ελεύθερη διακίνηση και διαμονή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εφαρμογή μιας απλούστερης διαδικασίας ψηφοφορίας, για παράδειγμα το e-voting, ώστε να αυξηθεί η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες και ειδικότερα στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να προσφύγουν στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή του κράτους μέλους που διαμένουν και τέλος την πρόθεση της αγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της χρήσης διαδικτυακών πλατφόρμων που πράγουν τις αξίες και τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα καταθέσουμε τις δικές μας Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Αν όχι, τότε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα και να προσθέσω ότι έως τις 12 του Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. 12 Οκτωβρίου, ξαναλέω, μέχρι τις 3 το απόγευμα. Και στις 21 Νοεμβρίου θα γίνει η ε, ψηφοφορία. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι από τη συζήτηση προκύπτει ότι όλοι έχουμε περίπου την ίδια κατεύθυνση ο στόχος είναι να κάνουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο να πιάνει τις βασικές σκέψεις που είναι η αποτελεσματικότητα ουσιαστικά γύρω από την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Εκ των πραγμάτων λόγω και των ευρωεκλογών δίνουμε μεγάλη έμφαση στα εκλογικά δικαιώματα αλλά βεβαίως με τις τροπολογίες φαντάζομαι και τις δικές σας και τις δικές μου θα καλύψουμε όλες τις πλευρές ούτως ώστε να έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις εκ μέρους των συναδέλφων και θα προετοιμαστούμε για τις τροπολογίες όπως είπατε μέχρι 12 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. για λόγους πληρότητας έχουμε, επί, έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ μαζί μας. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ακούμε. I'm Marine Boulanger. I'm head of unit in charge of EU citizenship rights and uh, I will be brief but welcome very much the opportunity. Πολύ σύντομα. Για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και σχετικά με τη γνωμοδότηση αυτή που μόλις παρουσιάσαμε που μόλις μας παρουσιάσε ο κ. Μαριάς. Ε, το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ε, αποδίδεται η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ιθαγένεια ε, αποδίδεται σε όλους τους πολίτες κρατών μελών. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την ελευθερική κυκλοφορία, την και που υπάρχουν και διατάξεις στην Τρίτη που υποχρεώνουν την Κομισιόν να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με την Ιθαγένεια. Και υπάρχει και ο συγγητής εδώ της Επιτροπής σχετικά με την έκθεση αυτή τη τελευταία της Κομισιόν και η συνθήκη επίσης προβλέπει και μια σειρά από άλλες διαδικασίες διεύρυνσης αυτής της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η Κομισιόν έχει λοιπόν ε, εκδώσει έκθεση πέρσι και θέλω να αναφέρω κάποια από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αλλά όσον αφορά την ελευθερή κυκλοφορία, η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση για το IDCAT και τα έγγραφα Διαμονή, κάτι που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, θα ενισχύσει και την ασφάλεια των εγγράφων αυτών που είναι πολύ σημαντικό για να αποφευθεί η απάτη και η παραποίηση και αυτό το εξετάζουν οι συνομοθέτες αυτή τη στιγμή, αυτή την πρόταση. Επίσης, προωθούμε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα. Έχουμε ε, εκδώσει και μια σχετική έκθεση για τις τοπικές εκλογές που θα γίνουν φέτος για τους ε, πολίτες που ζουν εκτός ε, του κράτους μέλους τους για την, την συμμετοχή τους στις τοπικές εκλογές. Δηλαδή έχουμε συντάξει έναν κατάλογο βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων και την προώθηση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο. Ε, κάναμε ένα εργαστήριο στο πλαίσιο το, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών κάποια project για αυτή τη βδομάδα ε, ε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Φέτος επίσης ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών διότι ε, τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, όπου και, το, την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών μάλλον σε τρίτες χώρες γιατί ξέρετε ότι είναι μια πολύ σημαντική οδηγία αυτή ε, για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους πολίτες ε, να την χάνουν της ε, προξενικής προστασίας, ε, της από τις προξενικές αρχές ε, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό και χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά έγγραφα. Εδώ μιλάμε για το ταξιδιωτικό έγγραφο έκτακτης ανάγκης. Επίσης, βρισκόμαστε σε στάδιο διαπραγμάτευσης ε, προσεγγίσεις προστασίας με τρίτες χώρες για να προστατευτούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών μας όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Αναφερθήκατε στα εκλογικά δικαιώματα ε, και στο δικαίωμα ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και εμείς θα εξασφαλίσουμε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες μας στην ιστοσελίδα μας εν των ευρωεκλογικών και βρισκόμαστε επίσης και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε, σε αντίστοιχες κινήσεις. Επίσης αναφερθήκατε στη σημασία της διαφάνειας. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει μια πολύ σημαντική σύσταση φέτος ε, στην δέσμη μέτρων για τις εκλογές και πολύ σημαντική ενέργεια ήταν και αυτό που έγινε πέρσι ε, σχετικά με την προστασία της ακαιρεότητας των εκλογών ε, την καταπολέμηση των ψευθών ειδήσεων. Έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη ε, την εφαρμογή αυτής της δέσμης μέτρων. Ε, φέτος, το Σώμα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που είναι ένα υψηλού επίπεδου σώμα εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξετάσει αυτά τα θέματα εν ώψη και των ευρωεκλογών. Να πω κάτι για το όριο και το e-voting Αυτά ε, αναφέρονται και στο νέο εκλογικό νόμο που, που ενέκρινε πρόσφατα το Συμβούλιο. Και για να κλείσω, θέλω να τονίσω ότι η προώθηση και η ανάπτυξη ευρωπαϊκής ηθαγένειας είναι κοινή αρμοδιότητα, ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όλων των θεσμικών οργάνων. Η Κομισιόν εκφράζει την προσήλωσή της στο να καταστεί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια μια πραγματικότητα και συνεργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με εθνικές τοπικές αρχές, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών ε, και με οργανώσεις πολιτών. Γιατί ε, λαμβάνουμε πολλές, ε, πολλές προφορίες και από τους ίδιους τους πολίτες γιατί πολύ συχνά λαμβάνουμε ερωτήματα από τους ίδιους πολίτες για το ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα ασκήσουν. Ευχαριστώ. Κύριε Μαριά, θέλετε το λόγο μια τελευταία φορά? Όχι. Εντάξει. Όπως είπα λοιπόν, Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου έχετε δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες. Ε, να δώσουμε όμως το λόγο και στον κύριο Αλεμάνη για να μας ξαναμιλήσει για το ζήτημα του οικοτόπου στο Πεγκολίβα. Παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά κύριε Αλεμάνη. Ωραία, θα είμαι σύντομος για να δώσω μια απάντηση πρώτα-πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να είναι γνωστά. Πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η έρευνα. Ε, γυρίζω να αφορά αυτή την ε, αστική περιοχή, όταν λέτε ότι δεν έχουμε σε αυτό το κυσκόσιο των 2000, άρα δεν συνιστά αυτό στην ναι, αλλά αυτή η περιοχή, το Μόντε Πέγο, υπάγεται ε, σε τρεις δήμους ντέμια, πεπέγο κλπ. Επομένως, νομίζω ότι εδώ είναι ανακριβή η ενημέρωσή σας. Εμείς ε, κατοικούμε σε ένα, ένα, ένα από τους τρεις αυτούς δήμους. Μιλάμε για πάνω από 4.000 συνολικά κατοίκους. Ε, και ε, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι το πέγο ε, συμμορφώνεται με την νομοθεσία όταν λέμε ότι δεν είναι ε, δεν είναι μόνο αυτός ο Δήμος που έχει το, τις εγκαταστάσεις καθαρισμού του ύδατος. Ε, είναι ένα κομμάτι μόνο. Το είπαν διάφοροι βουλευτές και συμφωνούν. Τώρα όσον αφορά την οδηγία για τον βιότοπο, είναι υποχρεωτικό τα κρατημέλη να ασκούν τη διαχείρισή του. Και στη σχετική οδηγία, στο άρθρο 4, ορίζεται ότι υπάρχει υποχέρωση διαδικασίας και προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους όποτε υπάρχει περίπτωση κινδύνου. Μα έχουμε ό,τι στοιχεία χρειάζονται για να καταλήξουμε στο ότι υπάρχει κίνδυνος. Πέραν από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουμε ένα σώρο ανεξάρτητους φορείς που το έχουν βεβαιώσει. Και τελευταίο, αυτές οι αναλύσεις που κάναμε στο φυσικό πάρκο αποδεικνύουν ότι όχι σε 450 ούτε σε 20 μέτρα. Είναι μέσα, μέσα ε, η μόλυνση από αυτά τα λίμματα. Αν δεν κάνουμε κάτι, τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Καταλαβαίνετε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας τα πω. Ο Πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Αλεμάνη. Υπενθυμίζω την απόφαση που λάβαμε. Ε, η ε, αναφορά παραμένει ανοιχτή και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε μελλοντική μας συνεδρίαση. Λοιπόν, αυτά και συνεχίζουμε αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 το πρωί. Καλό σας βράδυ.